Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ich erkläre die am zehn Mai das Protokoll und die angenommenen Texte der Sitzungen vom neun Τα πρακτικά τη 9 η και 10 η Μαΐου του 2012 είναι διαθέσιμα. Υπάρχουν κάποιε παρατηρήσει. Όχι. Θεωρώ λοιπόν ότι εγκρίνονται τα πρακτικά αυτά. Η κυρία Ντάβα Δευρούν με ενημέρωσε για την παρέτησή της από τις 3 Μαΐου του 2012 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το σημειώνουμε και σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού του Κοινοβουλίου είναι κενή η θέση της από την ημερομηνία αυτή. Οι αρχές της Ρουμανίας με ενημέρωσαν ότι η κυρία Μνοβάνα Πλούμπ θα αντικατασταθεί από τις 18 Μαΐου από την κυρία Μινόρντα Κλιβέτη. Καλωσορίζουμε λοιπόν αυτήν την νέα συνάδελφο, η οποία βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 2 μπορεί να